Α, ανακοινώσεις Προέδρου, δεν έχω όμω τέτοιε. Το δεύτερο είναι το 5Β, αποφάσει των συντονιστών, που έλαβαν δηλαδή στην ε, σημερινή πρωινή συνεδρίασή τους. Η πρώτη απόφαση των συντονιστών σήμερα το πρωί ήταν για θέματα ε, οικονομικών συμφερόντων των υποψηφίων ε, επιτρόπων Σίμψον και Πάσκου αποφάσισαν οι συντονιστέ να στείλουμε επιστολή στην διάσκεψη Προέδρων ε, Επιτροπών, διότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν αναλάβει χαρτοφυλάκιο και θεωρεί η Νομική Επιτροπή ότι δεν μπορεί να κρίνει για ζητήματα συγκρούσεως ε, οικονομικών συμφερόντων και θα αναβληθεί για την 3η Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη απόφαση των συντονιστών. Η δεύτερη απόφαση ήταν η κατανομή βαθμών στις πολιτικές ομάδες και όχι κατά βαθμών σε μη εγγεγραμμένους βουλευτές, οι οποίοι όμως μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία να γίνουν εισηγητέ, να λάβουν έκθεση δηλαδή και τότε θα ληφθεί απόφαση από τους συντονιστές αναπερίπτωση. Η τρίτη ε, απόφαση ήταν να λάβει, λάβει η Προεδρία της Νομικής Επιτροπής εντολή για να καταθέσει τροποποιήσεις ε, για, ε, στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε όνομα της Νομικής Επιτροπής και επίσης για τον αναπληρωτή διευθυντή του οργανισμού ή του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας πριν να ε, ορίσει το συμβολιο τον ε, επόμενο ε, αναπληρωτή διευθυντή και για διαρκείς εισηγητές μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Επομένως, ισότητα φύλων, S&D, παρατηρητής για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην ε, Χάγη Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Διαδικατικός διάλογος στην ομάδα Renew. Για πρόσωπα με αναπηρίες, διαρκή εισήγηση πράσινη. Επίσης το άλλο θέμα για τους αναπήρους. Και για το δίκτυο αναφορών στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να διαβιβάσουν λίστα με μη ολοκληρωμένε υποθέσει στην Προεδρία του Κοινοβουλίου για να ολοκληρωθούν οι, ε, οι υποθέσεις αυτές. Ο κύριο Δεμπλάνκο από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε για την άρση ασυλίας του βουλευτού Φερνάντε. Οι συντονιστέ, εγκρίνουν το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το 2020 και να ζητηθεί η έγκριση για διαμεθοριακές επιστροφές αποζημιώσεις ε, κλεμμένων αντικειμένων τέχνης. Οι συντονιστές συμφώνησαν επίσης να αποστείλουν προσκλήσεις και σε άλλες ε, συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτισμού. Στα δεύτερη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση για την βελτίωση της νομολογίας και για τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας και της ενίσχυσής τους στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου 2018 και για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού, της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι συντονιστές θα προσκαλέσουν επίσης εκπροσώπους για να καταθέσουν τι κατευθύνσει γραμμέ δεοντολογίας και συμφώνησαν επίση όπω και σε προηγούμενα χρόνια να ζητήσουν έγκριση για τις νέε εκθέσει, ετήσια έκθεση για την αναλογικότητα και επικουρικότητα, την παρακολούθηση τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου 2017 και 2018, αναθέτουν εντολή στη γραμματεία οι συντονιστέ πάντα να εξετάσουν θέματα κατευθύνων γραμμών και ε, ασυλιών. Οι συντονιστές αποφασίζουν να υποβάλουν προτάσεις στη γραμματεία για προτινόμενες συνεργασίες με εθνικά κοινοβούλια μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου. Αποφάσισαν επίσης να στείλουν προτάσεις για δημόσιες ακροάσεις για το δεύτερο εξάμεινο του 2019 πάλι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Αποφάσισαν επίσης επιγραπτής διαδικασίας η οποία θα διατυπωθεί κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών για τις, για τις επιταχυμένες διαδικασίες και θα τις υποβάλουν στην Επιτροπή μέχρι τέλος Ιουλίου. Αυτές ήταν όλες οι αποφάσεις. Ελπίζω να προλάβατε να τις καταλάβετε, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, ορίστε, ναι. Μα ενδιαφέρει πολύ η ακρόαση για τα κλεμμένα έργα τέχνης του Δεκεμβρίου. Είναι μεγάλη σημασία να συμμετάσχουμε στις ακρόασεις αυτές ως μέλη της Νομικής Επιτροπής. Αναμένω το πρόγραμμα, φαίνεται αρκετά ευρύ. Είμαι βεβαία ότι οι οργανωτές θα μπορέσουν να τα περιλάβουν όλα. Τώρα έχω μια ιδέα για μια συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια όπου η προθεσμία ήδη προβλέπεται μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, διότι αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μα να εξετάζει δηλαδή την επικουρικότητα, θα έχει ενδιαφέρον να γίνει κάποια συνεργασία με κάποιες εθνικές βουλές σχετικά με το πώς βλέπουν οι εθνικές αυτές βουλές την επικουρικότητα και ίσω με συμμετοχή γραμματιών των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Βουλών να μα προσεγγίσουν και να ανταλλάξουμε απόψει ενδεχομένω μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Αν συμφωνείτε και εσεί οι υπόλοιποι. Καλώ, θα τα συζητήσουμε αυτά μετά τη συνάντηση. Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο είναι το σημείο 6, το οποίο αναβάλλεται. Και περνάμε στο σημείο 7. Νομίζω εδώ πρόκειται για τον ορισμό του συγητή. Λοιπόν, κάποιες διορθώσεις σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Προβλέπεται γλωσσική εξέταση των πράξεων αυτών. Και ο σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι η διασφάλιση της ε, συνεκτικότητας με τις συνθήκες και με το σύνολο της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, με απλή γλώσσα τι σημαίνει αυτό, ότι τα νομικά έγγραφα έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει γίνει ο γλωσσικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός συνήθως γίνεται μετά τη πολιτική συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά πριν την έγκριση από την Ολομέλεια. Και όταν δεν υπάρχει ο χρόνος γι' αυτό, όπως για παράδειγμα στο τέλο τη ε, θητείας του Κοινοβουλίου, η πολιτική συμφωνία εγκρίνεται πρώτα στην Ολομέλεια και κατόπιν ε, διεξάγεται ο γλωσσικός έλεγχος. Το αποτέλεσμα έχει ήδη διαβιβαστεί και σύμφωνα με το άρθρο 231 του ιστορικού κανονισμού η Επιτροπή μας θα εξετάσει το τελικό κείμενο και θα καταθέσει το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια εφόσον είναι ικανοποιημένη. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλουμε το ε, διερθωμένο κείμενο στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Θα ήθελε κάποιος ε, το λόγο. Ωραία λοιπόν, δεν βλέπω αντίρρηση, μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε το κείμενο στην Ολομέλεια. Σημείο 8. Για να τηρηθούν οι προθεσμίες και σύμφωνα με την τακτική της Επιτροπής μας προτείνω να ε, κατατεθούν τροπολογίες επί του προϋπολογισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 20 Ιουλίου 2019. Οι τροπολογίες επί του προϋπολογισμού έχουν στόχο να ε, διορθώσουν τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου για ορισμένες ε, θέσεις προσωπικού οι οποίες έχουν περικοπεί από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Και δεδομένης της φύσης των θέσεων αυτών το Συμβούλιο προτείνει να επανέλθουν αυτές ε, οι θέσεις προσωπικού έτσι ώστε το δικαστήριο να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Να σας πενθυμίσω επίσης ότι το δικαστήριο σε αντίθεση με τα άλλα θεσμικά όργανα που είναι σε θέση να ελέγχουν το ε, το έργο τους δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων. Δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να απορρίπτει κάποια υπόθεση. Και έχει παρατηρηθεί λοιπόν μία αύξηση του φόρτου εργασίας κατά 80% μεταξύ 2012 και 2018. Η πρόταση λοιπόν επιστροφής ορισμένων κονδυλίων για τον προπολογισμό του 2020 ενέρχεται σε 440,6 ευρώ, ε, εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις. Φέτος λοιπόν ο προϋπολογισμός ε, θα δεχθεί διορθωτικές τροπολογίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή ε, Γιούρι, σε εμά δηλαδή. Προτείνονται λοιπόν ε, τροπολογίες που αφορούν τη δέουσα επιμέλεια, την ασφάλεια, τη, τα συστήματα πληροφορικής και θέματα προστασίας των καταναλωτών. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε για την εντολή unblock και να το κάνουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ήθελα, θα να πάρει το λόγο πριν προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Όχι. Ωραία λοιπόν. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Άρχεται. Ωραία λοιπόν, η πλειοψηφία είναι υπέρ της ε, χορηγής εντολής. Σας ευχαριστώ. Σημείο 9. Διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Όχι. Ωραία λοιπόν, προχωρούμε πολύ γρήγορα. Σημείο 10. Προσοχή συνεδριάσεις. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, θα έλεγε χώρα στις 3 Σεπτεμβρίου από τις 9 ως τις 12.30 και μετά από τις 2.30 ως τις 6.30.